Βαντεκάμπ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Βιμ Βαντεκάμπ. Έχετε το λόγο. Τέσσερα λεπτά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να μιλήσω απευθυνόμενο στους του ηγητέ, τους συναδέλφους για να τους ευχαριστήσω. Εκείνους όπως και κάθε άλλον που έλαβε μέρος σε αυτήν την ε, μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση. Θα ήθελα να απευθύνω τα πιο θερμά μου, τις πιο θερμές μου ευχαριστίες. Έχουμε πίσω μας αφήσει μια μακρά διαδικασία με 603 τροπολογίες. Μια διαδικασία επίπονη δεν ήταν εύκολο να καταλήξουμε σε ένα αφήγημα συνεπές. Και έτσι θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, της ομάδας μου αλλά και των άλλων ομάδων για τη συνεργασία. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό να το αναφέρω σχόλια για τις λευκές βίβλους καταρχάς. Οι πρώτες ήταν πολύ επιφυλακτικές, ε, λεγόταν ότι δεν υπάρχει πραγματικά νέα πολιτική, οι αποφάσεις δεν είναι πράγματι ενδιαφέρουσες και ουσιαστικές, αλλά νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε εδώ με μια μεσοπρόθεσμη μόνο αξιολόγηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση που παρουσιάζει κάθε τέσσερα χρόνια ε, μια νέα πολιτική δεν νομίζουμε ότι κάνει το βέλτιστο. Εμείς ζητούμε με την μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση πάνω απ' όλα μια συνέχεια στις πολιτικές. Στις κάτω χώρες έχουμε φτάσει να λέμε ότι πια δεν κινείται τίποτα. Ε, οι μεταφορές είναι πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Είναι ένας ε, τομέας που απασχολεί εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους, εκατομμύρια εργαζομένους. Δεν πρέπει να το μόνο με αυτό. Και αγαπητοί συναδελφοί, πρέπει να γίνει πιο βιώσιμος αυτός ο τομέας, το 25% των μεταφορο... Ε, της ε, ρήπανσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχεται από τις μεταφορές. 29% από το τομέα της ενέργειας, για να καταλάβετε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Η βιωσιμότητα λοιπόν, η, η αηφορία δεν μπορεί να θεωρηθεί όμως απειλή, αλλά ευκαιρία για καινοτομία στον χώρο των μεταφορών. Και θα πρέπει να επενδύσουμε σε αυτή την καινοτομία στις μεταφορές τα επόμενα 20-25 χρόνια. Ας κοιτάξουμε λοιπόν κάποια από τα σημεία της έκθεσης με τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση αυτή. Πρέπει καταρχάς να σημειώσουμε ότι η αλλαγή των επιλογών από το ένα είδος των μεταφορών σε άλλο, από τις οδικές και ενέργειες μεταφορές στο σιδηρόδρομο και τις εσωτερικές πλωτές οδούς, δεν έχει υλοποιηθεί. Παρότι θέλουμε να έχουμε πιο καθαρές μεταφορές, πράγμα που εξασφαλίζουν οι συνδρομικές και πλωτές μεταφορές, δεν έχει αλλάξει η επιλογή. Πρέπει λοιπόν να προωθηθούν οι συνδρομικές μεταφορές και οι εσωτερικές πλωτές και θαλάσσιες μεταφορές. Σε αυτό συμφωνούμε. Ε, τα ευφύ συστήματα μεταφορών επίσης, Πρόεδρε, ITS. Σε αυτά θέλουμε περισσότερη καινοτομία. Πρέπει να τα έχουμε εξασφαλίσει τα συστήματα αυτά σε πλήρη λειτουργία στο 2020. Το θέμα που αφορά τις ε, αστικές μεταφορές θα το εκθέσουν οι συνάδελφοι ασφαλώς. Ε, ίσως να έχω λίγο περισσότερο χρόνο. Μάλλον όχι. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Σιγητά και εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής η κυρία Βιολέτα Βούλτς έχει το λόγο. Πρόεδρε, ε, αγαπητοί ε, ευρωβουλευτές, θα ήθελα να, τον, να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τους ε, σκιώδους αλλά και όλο το Κοινοβούλιο για την πολύ χρήσιμη ε, συνεργασία στην εφαρμογή της Λευκής Βίβλου. Πάνω από 600 τροπολογίες ε, υποβλήθηκαν και αυτό αποδεικνύει το ενδιαφέρον που δημιουργεί το θέμα στους ευρωβουλευτές. Η Κομισιόν Ιεκά είναι ικανοποιημένη με το περιεχόμενο και την κατεύθυνση που ακολουθεί η έκθεση. Θέλω όμως να σχολιάσω 7 συγκεκριμένα σημεία. Πρώτον, ε, η πρόθεση των πολυτροπικών ε, μεταφορών στηρίζουμε αυτό το στόχο. Γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες, να εσωτερικοποιήσουμε τα εξωτερικά κόστη, να συμπληρώσουμε ε, τις απουσίες υποδομών, να αντιμετωπίσουμε θέματα διαλειτουργικότητας και να διασφαλίσουμε υγιή ανταγωνισμό μεταξύ όλων των μέσων. Δεύτερον, συγχρονισμός της ε, υποδομής. Εδώ έχουμε σημαντική πρόοδο πλευράς Κομισιόν ο ορισμός των διαδρόμων των διευρωπαϊκών δικτύων και ο μηχανισμός ε, συνέοντας στην Ευρώπη ήταν από τα βασικά βήματα που κάναμε τα τελευταία χρόνια. Πολλά project θα μπορέσουν να χρηματοδοθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων. Τρίτον, η βιωσιμότητα των μεταφορών. Εδώ είναι μια περιοχή στην οποία η Κομισιόν θα παραμείνει πολύ δραστήρια. Ε, μείωση της χρήσης του άνθρακα αλλά και ε, μείωση της ε, χορύπανσης, νοσφαιρικής ρήπανσης κλπ. οι νέε μεταφορέ θα πρέπει να ψαχθούν ιδιαίτερα, αλλά να προσέξουμε έτσι ώστε οι λύσει μα οι λύσει που θα προτείνουμε να είναι ρεαλιστικέ. Τέταρτον, οι ψηφιακέ λύσει συμφωνούμε ότι πρέπει να βελτιώσουμε τις πληροφορίες για, τις, ε, για τα ταξίδια και να ε, δημιουργήσουμε ολοκληρωμένα συστήματα ε, διαχείρισης εισιτηρίων. Όμως δεν είναι δυνατόν να επιβληθεί μία λύση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει οι πληροφορίες να είναι διαθέσιμες και οι εταιρείε ας βρουν τις λύσεις που θα ταιριάζουν στους πελάτες τους. Εμείς θα αναπτύξουμε πρότυπα και κανονιστικά πλαίσια έτσι ώστε να βοηθήσουμε καινούριε ε, υπηρεσίες να αναπτυχθούν, υπηρεσίες προσθέμενης αξίας. Η έκθεσή σας επίσης σχετίζεται και με το πέμπτο σημείο, ε, ο άνθρωπος να μπει στο κέντρο, στο επίκεντρο της πολιτικής μεταφορών μας. Συμφωνώ απόλυτα. Προσωπικά πιστεύω ότι οι μεταφορές θα πρέπει καταρχήν και κυρίως να ε, ωφελεί την κοινωνία τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τη μεταφορά αγαθών κλπ. Έκτον, κοινωνικά ζητήματα. Η σημερινή κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική. Η Επιτροπή Juncker αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο να αντιμετωπίσει το θέματα των ανεπαρκών συνθήκων εργασίας, ανεπαρκών προσόντων κλπ. Ε, μόνο με τέτοιου είδους μέτρα θα βελτιώσουμε την εσωτερική αγορά μεταφορών. Έβδομον, πιο αποτελεσματικέ και ανταγωνιστικέ μεταφορές και εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικοί φραγμοί στην Ευρώπη που επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία της ενίας αγοράς μεταφορών. Σταδιακά προσπαθούμε να καταργήσουμε αυτούς τους φραγμούς και να δημιουργήσουμε μια ενία ευρωπαϊκή ε, ε, αγορά μεταφορών Κάτι που θα επιτρέψει την Ευρώπη να παραμείνει ηγέτιδα στον τομέα των μεταφορών στον κόσμο. Τέλος, υπογραμμίζει η εκθέση σα ότι μία από τις βασικές αδυναμίες τη σημερινή των σημερινών μα πολιτικών είναι ε, η ανεπαρκής εφαρμογή. Συμφωνώ απόλυτα. Και νομίζω ότι εδώ θα μπορούσαμε ενδεχομένω να συνεργαστούμε πιο στενά έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ιδιαίτερα ότι η κοινωνική νομοθεσία θα είναι όσο πιο σαφής και αποτελεσματική γίνεται και ώστε να ε, ε, γίνουν ε, προσπάθειες χρειάζονται προκειμένου να εφαρμόζεται σωστά. Ε, η δουλειά μας είναι μακρόπνοη και αναμένω ότι θα συνεργαστούμε και στο μέλλον με έναν τρόπο βιώσιμο και επικοδομητικό καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Και τώρα... Εκ μέρους των πολιτικών ομάδων οι επόμενοι ομιλητές, καταρχάς εκ μέρους του ΕΛΚ, ο Μάρκος Πίπερ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η έκθεση προσφέρει πολλές καλές ενδείξεις για μια πιο ισχυρή διαλειτουργική διασύνδεση αηφορία στις μεταφορές και διασυνοριακές μεταφορές. Θεωρητικά όλα αυτά ακούγονται πολύ ωραία. Ωστόσο κύριε και κύριοι, το χώρο των μεταφορών, το μέσο των μεταφορών έχει ένα ιδιάζον χαρακτηριστικό αυτή τη στιγμή πολιτικά. Είναι ε, μια γαλακτοφόρος αγελάδα της Ευρώπης. Α, υποχρεούται όλο και περισσότερο να ε, τηρεί αυστηρές ε, προδιαγραφές για το περιβάλλον, επιβάλλονται όλο και πιο πολλές ρυθμίσεις, ρυθμίσεις όχι μόνο στα οικονομικά, μεταφέρονται όλο και περισσότεροι ε, επιβάτες. Και τα στοιχεία έχουν να κάνουν με φόρους διαφόρων ειδών που επιβάλλονται από τα κράτη-μέλη σε σχέση με την ε, προστασία του περιβάλλοντος ε, ή τα έσοδα των κρατών. Και πρέπει να ρωτήσω γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να λάβει τα χρήματα από την ε, διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη για να χρηματοδοτήσει πράγματα τα οποία δεν ήταν σχετικά. Λυπούμε που το ρωτώ. Έχουμε πολύ κακή ε, χρηματοδότηση των διεθνικών, των υπερσυνοριακών ε, μεταφορών, των υποδομών των μεταφορών και έχουμε να κάνουμε μια σειρά από προβλήματα τα οποία φαίνεται να προβάλλουν ε, ως, από τα οποία φαίνεται να προβάλλεται το ποδήλατο ως λύση για τις μεταφορές. Χρειάζεται διαφορετικές λύσεις ο χώρος των μεταφορών. Ο κύριος Φαντανκάμπ κατά εξαιρετικό τρόπο τα περιγράφει Θέλουμε και αηφορία και ανταγωνιστικότητα και υποδομές και επιχειρήσεις που θα δρουν αποτελεσματικά για να μην χάσουμε τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, τον παγκόσμιο αγώνα της ανταγωνιστικότητας. Σας ευχαριστώ. Ε, εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η κυρία Ταπαρτέλα. οσκι Κύριος Λοτόφσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν ενιαίο χώρο μεταφορών στην Ευρώπη, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι πρόκειται για κάτι δύσκολο και προκειμένου να επιτύχουμε πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης, θα πρέπει να καθορίσουμε την κατάσταση και τους ευρύτερους στόχους μας. Η Λευκή Βίβλος για τις μεταφορές είναι αυτό το σχέδιο, αυτή είναι η φιλοδοξία μας. Αλλά εγκρίναμε αυτή τη στρατηγική ε, πριν από τέσσερα χρόνια Παρά το γεγονό αυτό, διαπιστώνουμε ήδη ότι υπάρχει μια καθυστέρηση όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων. Κάποιοι από αυτού του στόχου δεν ήταν ρεαλιστικοί και ήταν εξαιρετικά ε, φιλόδοξοι. Παραδείγματο χάρη, ε, να μην υπάρχει καθόλου χρήση ορυκτών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών. Αυτό ήταν ένα πολύ φιλόδοξο όραμα. Τώρα γίνεται μια αναθεώρηση τη Λευκής Βίβλου. Πρέπει λοιπόν με αυτή την ευκαιρία να επικεντρωθούμε στου ρεαλιστικού στόχου. Η ολοκλήρωση του τομέα των μεταφορών είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συμβεί επί τόπου. Θα πρέπει να επισημάνουμε τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Προγράμματα όπως το πρόγραμμα των διευρικών δικτυαίων είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να ενισχύσουμε την ολοκλήρωση του τομέα των μεταφορών και αν θέλουμε να υπάρχουν ε, διαθέσιμες, ε, ε, διαθέσιμε μεταφορικά μέσα σε απομακρυσμένες περιοχές, τότε θα πρέπει να είναι προτεραιότητα οι μεταφορές στις πολιτικές μας στα επόμενα χρόνια. Η Λευκή Βίβλος ως έχει δεν αναφέρεται παρκώς ε, στην αστική κινητικότητα και στις αστικές μεταφορές. Δεν αναφέρεται παρκώς ε, στην, ε, στη μορφή car sharing και άλλες αντίστοιχες μορφές συνεργασίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το έγγραφο και αυτά τα ζητήματα δεν πρέπει να παραγνωρίζονται. Αν θέλουμε επίση να μιλούμε για το μέλλον του τομέα των μεταφορών, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε και του εργαζομένου του τομέα κάποια κράτη-μέλη προσπαθούν να προστατεύσουν τους επιχειρηματίες τους εις βάρος των οικονομικών ελευθεριών που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την αιτιολογία τη... Ε, κοινωνικού κόστους. Ε, χαίρομαι λοιπόν που ο εισηγητής αναφέρεται στην κατάλληλη ισορροπία μεταξύ εσωτερικής αγοράς και προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ελπίζω να τίνει ευήκονους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να λάβει υπόψη της και το σχόλιο αυτό και πολλά άλλα σχόλια τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση για να μπορέσουμε να έχουμε και κατάλληλη εφαρμογή της. Ευχαριστώ. Ε, Κυρία Ταπαρδέλ. Κυρία Ταπαρδέλ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η παγκοσμιοποίηση, η αστιφιλία, οι δημοκρατικές αλλαγές στις κοινωνίες μας μας, κάνουν να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που λειτουργούν οι μεταφορές. Διαπραγματευθήκαμε μια φιλόδοξη ατζέντα μέσω της Λευκής Βίβλου πριν από τέσσερα χρόνια με στόχο να δημιουργηθεί μια, ένα ενίος χώρος μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες των επιβατών και της μεταφοράς φορτίων τον 21ο αιώνα και να βοηθήσει την κινητικότητα. Για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να μπει στο κέντρο των συζητησιών μας ο επιβάτης. Θα πρέπει να ε, καθορίσουμε ελάχιστες προδιαγραφές για το κάθε μέσο μεταφοράς. Σε ό,τι αφορά την νέα αγορά θα πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή της, των ίσων ευκαιριών. Και επίσης θα πρέπει ο τομέας των μεταφορών να γίνει πιο ελκυστικός για τις γυναίκες. Θα πρέπει να καταργηθούν οι φραγμοί και να χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα μεταφοράς με βιώσιμο τρόπο. Χρειαζόμαστε και υλικές μεταφορές και, και ηλικιακές υποδομές και ψηφιακές υποδομές. Θα πρέπει να εστιάσουμε στην διασύνδεση των συνοριακών και των περιφερειακών περιοχών με όλες τις υπόλοιπες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε οι επιβάτες, φορτία και υπηρεσίες να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα και αποτελεσματικά. Χρειάζεται να γίνουν επενδύσεις σε αυτές τις περιοχές, δηλαδή παραμεθόριες και περιφερειακές περιοχές ε, και αυτές οι επενδύσεις θα επηρεάσουν πολύ και την ε, συνοχή, κοινωνική και οικονομική συνοχή. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μεταφορές στις πόλεις όπου παρατηρείται το φαινόμενο της αστιφιλίας. Εκεί οι μεταφορές αποκτούν ένα αρνητικό πρόσωπο πολύ συχνά. Ε, λόγω των συμφορήσεων, της μόλις του περιβάλλοντος, της χορύπανσης κλπ. Οι πληροφορία σε πραγματικό χρόνο και η χρήση της τεχνολογίας θα μπορούσε να μας βοηθήσει να λύσουμε τέτοια προβλήματα. Η μεταφορές ε, αποτελούν κινητήριο δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και θα βοηθάνε ακόμα και στην αύξηση του τουρισμού, για παράδειγμα, καθώς επίσης και στην βελτίωση των υπηρεσιών στους επιβάτες. Ε, behalf... Ευχαριστώ Ευχαριστώ εκ μέρους της ομάδας των Φιλελευθέρων, η κυρία Μάισνερ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συναδελφοί, κυρία Επίτροπε. Όντως, οι μεταφορές ε, δεν έχουν αξιολογηθεί σε, όλους τους, σε όλη τους την αξία. Ακόμα και αν δεν λειτουργούν σε, όλα τους τα, σε όλους τους τομείς, αποτελούν ραχοκοκαλιά της εσωτερικής αγοράς. Αν διανοηθούμε ότι μπορούμε να παραγγείλουμε κάτι στο ίντερνετ και να μας παραδοθεί μέσα 24 ώρες χωρίς μεταφορές, δεν γίνεται αυτό δεν γίνεται δυνατόν, ε, ε, η αποκομιδή των σκουπιδιών, ε, το να πάμε να δουλέψουμε σε ένα άλλο τόπο, τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς μεταφορές. Για τον πόλεμο χρειαζόμαστε καλές μεταφορές και γι' αυτό ο σχεδιασμός για τα υπόγειους σιδηροδρόμους στο μετρό δηλαδή ε, στην προηγούμενη χρονική περίοδο για όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ευρώπης ε, το, και το μεγάλο αυτό δίκτυο TNT είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό πρέπει να γίνεται χωρίς ε, εμπόδια, χωρίς περιορισμούς. Όλα αυτά λοιπόν είναι σωστά και καλά και χρειάζεται η κινητικότητα για τον πολίτη και τη μεταφορά των εμπορευμάτων για κάθε τύπου μεταφορά. Χρειαζόμαστε κάθε τύπου μεταφορές λοιπόν, ε, χρειαζόμαστε τους δρόμους, ε, τις ε, οδικές μεταφορές για τα εμπορεύματα, τις εσωτερικές πλωτές οδούς, θαλάσσιες οδούς, ακόμα και το ποδήλατο βεβαίως. Και αυτό πρέπει να γίνει κατά τρόπο οικονομικό, περιβαλλοντικό, ισότιμο για τον κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως των δυσκολιών που μπορεί να έχει λόγω μιας αναπηρίας, ε, με όρους ε, θεμητού ανταγωνισμού και βέβαια καλές συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους, αλλά και δικαιώματα για τους ε, επιβάτες. Όλα αυτά λοιπόν τα βλέπουμε μέσα στη μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση που μας λέει ότι πολλά πράγματα χρειάζονται ακόμα βελτίωση. Αλλά η βελτίωση θα πρέπει να προχωρήσει κατά τρόπο ισορροπημένο για όλους τους τομείς, για το χρήστη και για τον πάροχο της υπηρεσίας και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε προβλήματα όπως αυτά του Γιβραλτάρ που αποτελεί το μήλο τη έρηδα μεταξύ τη ε, Βρετανία και τη Ισπανία. Πρέπει να βρούμε για τι ενέργειε μεταφορέ ιδιαίτερα ε, μία λύση και στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρου τη ομάδα Γκουέντζιελ. Η κυρία Μαρία Κούλλορεν. arvoisa puhemies, komission jäsen. Επίτροπε, Ευχαριστώ πολύ στον κύριο Βαντενκάπ για την πολύ επικοδομητική του δουλειά. Είναι σημαντικό το έγγραφο αυτό για την Επιτροπή Μεταφορών. Η τελική του μορφή θα αντικατοπτρίζει και το όραμα μας για την πολιτική μεταφορών. Αναρωτιέμαι όμως αν έχει ληφθεί υπόψη επαρκώς η φωνή του καταναλωτή, του, η φωνή του πελάτη. Φαίνεται μερικές φορές σαν η, Επιτροπή η ε, πολιτική μεταφορών να είναι εκεί ώστε να διασφαλίσει τα συμφέροντα μόνο ε, των επιχειρηματιών ή των ε, εταιριών. Μερικές φορές σαν να ξεχνάμε τους πελάτες, τους επιβάτες. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι υποδομές είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι. Το πιο σημαντικό είναι τι γίνεται πάνω στις μεταφορές. Χρειαζόμαστε ευφυείς λύσεις και είναι κρίμα που ε, ναι, τη 2015 είναι πιο εύκολο να δημιουργήσουμε να χτίσουμε ένα αυτοκινητόδρομο μέσα από ένα βουνό, από το να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο, κανονιστικό πλαίσιο που θα βελτιώνει τις υπηρεσίες προσφέροντας τους πολίτες. Ε, ε, μερικές ε, φορές θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε πιο πολύ το καταστροφή εγγράφων παρά το μετροπόντικα. Ευχαριστώ. On behalf, Greens. Ευχαριστώ εκ μέρους των Πρασίνων. Ο Μπάς Άικχουτ. μισή λεπτό. Παρακαλώ. Ε, εντάξει, καλά είναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον συνάδελφο Βιμ Βαντεκάμπ, θερμά για τη συνεργασία. Θέλαμε ένα συμβιβασμό, αλλά δεν θέλαμε να είναι ένα κενό συμβιβασμό. Θέλαμε να υπάρχουν και κάποια στοιχεία μέσα σε αυτό και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βαντεγκάμ διότι ε, μπορεί με να μην έγινε πράσινο το κείμενο παντού, διότι δεν υπάρχει κατάλληλη πλειοψηφία, αλλά υπάρχουν αρκετά σημεία στα οποία ε, συμφωνούμε. Θα ήθελα να πω στην Επίτροπο ότι θεωρώ ότι είναι θετικό το γεγονό ότι αποδέχεστε την έκθεση, αλλά υπάρχουν αρκετά στοιχεία που χρήζουν βελτίωση. Αν δείτε την παρούσα κατάσταση των μεταφορών, το έθεσε και ο κύριος Βαντεκάπ, η μεταφορά ε, στις εσωτερικές ε, ε, πλωτές οδούς καθυστερεί, για παράδειγμα. Αν εξετάσετε το θέμα της μείωσης των εκπομπών και της ρήπανσης στις μεταφορές, ακόμα δεν έχουμε επιτύχει το στόχο μας. Πρέπει να επιτύχουμε τους στόχους μας πέρα από το 2020 και πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας προς αυτό το σκοπό. Χαίρομαι που έχουν συμπεριληφθεί και οικονομικά ζητήματα, αλλά το άνοιγμα προ την αγορά έχει και κάποιε προποθέσει. και θέλουμε και κάποιε δεσμεύσει και κάποια πρόοδο. Τα έχετε επισημάνει τα προβλήματα μεν, αλλά χρειαζόμαστε κάτι πιο συγκεκριμένο και είναι πολύ σημαντικό να θεωρήσουμε ότι η έκθεση αυτή αποτελεί ε, ένα κόδωνα κινδύνου προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι εναγκαλίζουμε προς τα μέτρα. Χρειαζόμαστε νέα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι μέχρι το τέλο τη περίοδου τη Λευκή Βίφλου θα είμαστε καθοδόν στην επίτευξη των στόχων μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λούγκρεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πριν από ένα χρόνο ανέλαβα καθήκοντα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αμέσως ε, άκουσα για τα προβλήματα που αφορούν τις μεταφορές. Πρέπει η νομοθεσία όμως να μας επιτρέπει να λαμβάνουμε μέτρα. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει μία εκ των υστέρων αξιολόγηση, κάτι το οποίο μας χαροποιεί μεν, ε, χαροποιεί και τους κατοίκους της χώρας μου που διοργάνωσαν και μια συγκεκριμένη διαδήλωση επί του ζητήματος. Ε, επιτέλους αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν προβλήματα και είμαστε διαδεθειμένοι να τροποποιήσουμε την νομοθεσία. Πρέπει να ε, καλύψουμε και τα κοινωνικά ζητήματα για να μην υπάρχει dumping στους μισθούς και να μην υπάρχουν ανισότητες ε, στους μισθούς. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε και τα παράνομα μέτρα, όπως για παράδειγμα το dumping στη μισθοδοσία. Θα θέλαμε να γίνει επιτέλους κάτι, ώστε να υπάρχουν ίσοι όροι ε, στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. η κυρία Αρνετού. Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθύτατη διαφωνία μου ως προς τις ε, προτάσεις εκθέσεως με πρόσχημα την καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Αυτή η έκθεση πάνω απ' όλα προσπαθεί να ενισχύσει την επικυριαρχία της Ευρωπαϊκής ε, Γραφειοκρατίας εις βάρος των κρατών μελών. Λυπούμε ιδιαίτερος για την, για την αύξηση των πόρων που ζητεί αυτή η Λευκή Βίβλος, που βεβαίως θα πρέπει να επιβαρύνουν τους φορολογούμενους των κρατών μελών και δι' τους Γάλλους. Ιδιαίτερα θα ήθελα να αναφερθώ στο χώρο του ανταγωνισμού, στο άνοιγμα του ανταγωνισμού, στους σειροδρόμους που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση εν τέλει. Είναι πολύ δύσκολο να δεχθούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τολμάει να υπαγορέψει στα κράτη-μέλη ε, όρους για την οδική ασφάλεια που περιορίζουν όλο και περισσότερο τις ελευθερίες για τα επόμενα χρόνια. Και όπως καταλαβαίνετε θα καταψηφίσω την έκθεση. Ε, Σας ευχαριστώ. Και τώρα... Ο κύριος Λουίς Δεγκράντες Πασκουάλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ, αξιότιμη συνάδελφη. Η πολιτική μεταφορών είναι σημαντικό στοιχείο της εσωτερικής αγοράς. Η, χωρική, η εδαφική συχνότητα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται από αυτήν. Ε, είναι πολύ σημαντικά τα δίκτυα μεταφορών, ιδιαίτερα στα μεθοριακά. Ε, είναι απαραίτητες οι μεταφορές για τον υγιή ανταγωνισμό και για την καθημερινή ζωή. Υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία στην έκθεση αυτή που θα ψηφίσουμε αύριο. Για παράδειγμα, εσωτερικοποίηση εξωτερικού κόστου, ε, αποφυγή διπλή φορολόγηση, εναλλακτικά κάψιμα, μέτρα για τι ε, μεταφορέ, το συνεπιβατισμό, ε, όλα όροι εργασία και συνθήκε εργασίας των μεταφορέων, ο ρόλος των μεταφορών στις ε, περιφερειακές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Ο εισηγητής έκανε πολύ καλή δουλειά και σίγουρα η ψήφος αύριο θα είναι θετική. Ένα όμως, μία μόνο αντίρρηση έχω να φέρω. Η αναφορά στο αεροδρόμιο του Γιβλαρτάρ δεν με βρίσκει σύμφωνο ως Ισπανό. Ποτέ δεν έχουμε μπλοκάρει το θέμα των μεταφορών ε, εξαιτία του Γιβλαρτάρ. Πάντοτε προσπαθούμε να βρούμε μια φιλική λύση μεταξύ δύο φιλικών χωρών, Ισπανία και Ενωμένο Βασίλειο οι κανόνες, ε, η, μάλλον η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί όταν ξεπεραστούν τα προβλήματα και η λύση θα βρεθεί μόνο μέσω του διαλόγου. Είναι ο μόνος δρόμος. Ε, δεν είναι λύση να λαμβάνονται τέτοιου είδους αποφάσεις από το Συμβούλιο γιατί άλλωστε δεν είναι και αρμοδιότητά του. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ Ισμαϊλ Αρτούχ. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμη Πρόεδρο, αξιότιμη, αξιότιμη κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς οφείλω ευχαριστήσω τους πρωταγωνιστές τον κύριο Φανανκάπ, εισηγητή, και την κυρία Ταπαρντέλη, τη δική μας και όδηση για την πολύ καλή δουλειά. Ήταν όντω για πολλές εβδομάδες μια πολύ καλή και επικοδομητική αυτή η συνεργασία και συγκινησιακά φορτισμένος ο διάλογος. Θα ήθελα να σημειώσω για άλλη μια φορά τη Λευκή Βίβλο που υιοθετήσαμε πριν από τέσσερα χρόνια. Πολλά ήταν τα φιλόδοξα μέτρα που είχαμε προτείνει. Βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο λοιπόν, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο τέρμα. κυριω όσον αφορά την μετατόπιση του βαρου των μεταφορών από τι οδικές στο σιδηρόδρομο, κυριω για τι μεταφορέ φορτίων άνω των 300 χιλιόμετρων. Αυτό δεν το καταφέραμε. Κινούμαστε σε ένα χαμηλότερο επίπεδο από το 2008 στο 2011 είχαμε ένα μέσο όρο των ε, εμπορευμάτων ε, που μεταφέρονται οδικός στο 67%. Ε, από την στην περίοδο 2011-2013 το ποσοστό αυτό έφτασε στο 74,3%. Ανωδική τάση λοιπόν, αλλά όχι ακόμη επαρκής όπως θα θέλαμε. Στον κοινωνικό τομέα επίσης πρέπει και θα ήθελα να παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τίνει χείρα προς το συνεργασίας προς το Κοινοβούλιο. Ε, στον κοινωνικό λοιπόν τομέα, στην ασφάλεια, έχουμε θέσει το δάκτυλο επί το τύπο των Ήλων και ζητούμε μέτρα συγκεκριμένα για τη βελτίωση της κατάστασης. Όσον αφορά τους επιμέρους τομείς, το pay to fly, το, την εικονική αυτοαπασχόληση και διάφορους άλλους τομείς πρέπει να δουλέψουμε ακόμη περισσότερο για να έχουμε αποτελέσματα. Κλείνοντας, κυρία Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ για την άτεγκτη ε, στάση σας στο θέμα του, ε, των διοδίων για τη Γερμανία. Ήταν πολύ ορθή η στάση σας και ελπίζω να έχουμε στο μέλλον πάλι τέτοια συμπεριφορά. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα η κυρία Τζάκλιν Φώστερ για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Φαντενκάπ για την πολύ σκληρή δουλειά του. Για μας είναι κρίμα για μας συντηρητικούς ότι άλλαξε μεγάλο κομμάτι του αρχικού σας κειμένου. Εμείς το υποστηρίζαμε, όπως ξέρετε. Κάποιους, κάποιες παραγράφους με δυσκολία θα δεν θα μπορούσε να τις υποστηρίξει η ε, αντιπροσωπεία των Βρετανών συντηρητικών. Υπάρχει κίνδυνος να ε, επηρεαστούν οι αγορές με προστατευτικά μέτρα, ιδιαίτερα όσον αφορά τις οδικές μεταφορές φορτίων. Το θέμα της υπηρεσίας για, για την ασφάλεια των μεταφορών δεν μας πείθει, δεν νομίζω ότι θα προσθέσει τίποτα. Η οδηγία για τους λιμένες όπως έχει μπορεί να είναι επιβλαβής για τα συμφέροντα της πολύ του πολύ επιτυχημένου κλάδου των Βρετανικών λιμένων και κλείνοντας θέλω αναφερθώ στο Γιβραλτάρ ο φίλος, που είχε, φίλος και συνάδελφος που είχε πριν από δύο χρόνια καταθέσει σχετικές τροπολογίες για αποχωρήσει από ό,τι βλέπω ξέρετε ότι πρόκειται για εδαφικό για τμήμα για έδαφο τη Βρετανία, όπου έχει κυριαρχικά δικαιώματα η Βρετανία, δεν αλλάζει αυτό. Στο θέμα των ενιαίων εθέρων ε, και ο κύριο Μπάχτο έχει επεξεργαστεί. Ε, δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει τίποτα και αυτός είναι ο λόγος κύριε Φαντενκάπ και αυτός είναι ο μόνος σοβαρός λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε την έκθεση σας ε, και τι εκτιμούμε πολύ τη σκληρή δουλειά σας γι' αυτόν και μόνο τον λόγο δεν θα μπορέσουμε να την υπερψηφίσουμε ελπίζουμε να κατανοείτε Σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος Και τώρα η κυρία Παλώμα Λόπεθ Μπερμέχο Ναι, ευχαριστώ πολύ και κυρίως ε, γιατί προφέρετε σωστά το όνομά μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε οι οδικές μεταφορές βρίσκονται σε μια μεταβατική περίοδο ε, εν αναμονή της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Το αίτημα για λειτουργικότητα, για περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα και την ανάγκη να έχουμε κοινού, από κοινού παραγωγή και διανομή στην Ευρώπη μας υποχρεώνουν να έχουμε ένα μοντέλο το οποίο εξαρτάται πάρα πολύ από τις μεγάλες υποδομές και τις μεγάλες επιχειρήσεις των μεταφορών. Σε αυτή τη ε, μεταβατική φάση είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεθεί στο επίκεντρο τη συζήτηση τα δικαιώματα και τα αιτήματα των εργαζομένων ε, και των αυτοαποσχολούμενων. Ε, θα πρέπει να δώσουμε μάχη κατά του κοινωνικού ντάμπινγκ. Ε, τα η κατάκριση των κανόνων του καποτάζ και των αποσπασμένων εργαζομένων είναι μια υπόθεση που σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν κατάλληλοι και πιο αυστηροί έλεγχοι και μια, υπάρχει σε ευθύνη του εργοδότη ή του υπεργολάβου. Ε, είναι απαράδεκτο να απελευθερώνεται ένα τομέα με μόνο στόχο να μην υπάρχει προστασία στι ε, συλλογικές και στους εθνικούς ε, κανονισμούς. Ε, θα πρέπει να κάνουμε κάτι καλύτερο γι' αυτό. Ευχαριστώ η κυρία Ντανιέλα Γιούτο τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρώ ότι έγινε εξαιρετική δουλειά στη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές, ε, την οποία όμως δεν υποστηρίξουμε ως αντιπροσωπεία των πέντε αστέρων, γιατί δεν θέλουμε να υποστηρίξουμε ε, έργα όπως ε, το, το Ρήνο Λιών, παρά το γεγονός ότι έχει αποδειχθεί ότι είναι επιζήμιο το έργο αυτό. Ε, και ε, παρόλα αυτά επιλέγεται να υλοποιηθεί. Προσπαθήσαμε με τροπολογία μας να βοηθήσουμε, όπως για παράδειγμα για να επενδύουμε σε βιώσιμες μεταφορές και να είμαστε υπέρ των σιδηροδρομικών μεταφορών και όχι των οδικών μεταφορών. Να προωθούμε τα ανακυκλούμενα μέσα, τα ηλεκτρικά μέσα, το car sharing, τη δημιουργία νέων σχεδίων αστικής κινητικότητας για να δώσουμε κίνητρα για τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και επίσης ε, να δώσουμε και μέτρα ε, κατά του κοινωνικού ντάμπινγκ. Παρόλα αυτά πρέπει να πω ότι είμαι αντίθετη στο κείμενο το οποίο εγκρίνθηκε. Για άλλη μια φορά θέλετε να δώσετε μεγαλύτερες εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να χρηματοδοτήσετε άχρηστα έργα τα οποία ε, είναι προς όφελος μόνο της Ευρωπαϊκής Ολιγαρχίας και των μεγάλων εξουσιών. Εξακολουθείτε να κάνετε λανθασμένες επιλογές για να μην παραδειχθείτε τα σφάλματά σα, όπως κάνετε και με το ευρώ. Ξέρετε ότι δεν έχει αποτέλεσμα αλλά συνεχίζετε συνεχίζετε με τι παράλογες πολιτικέ σα για να προστατεύετε την Ευρωζώνη. Κάντε σαν του αλκοολικούς, παρά το γεγονό ότι ξέρουν ότι θα πεθάνουν, πίνουν κονιάκ ακόμα και για πρωινό. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ. Κύριε Λουκατσέφσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι μεταφορές ε, είναι η ραχοκοκαλιά οποιασδήποτε οικονομία. Η εσωτερική αγορά δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς ε, σύγχρονες ε, μεταφορικές υποδομές. Θα πρέπει ο, των μεταφορών να μετασχηματιστεί, θα πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματικός, ε, πιο αποδοτικός ενεργειακά, πιο διαλειτουργικός. Οι στατιστικές δείχνουν ότι οι μεταφορές θα γίνονται όλο πιο αναγκαίες, η ζήτηση θα διπλασιαστεί. Συγχαρητήρια στον εισηγητή, εξαιρετική έκθεση με πολύ σημαντικά σχόλια για πολλά ζητήματα. Προφανώ, τα όσα προτείνουμε δεν αποτελούν πανάκια. Οι μεταφορέ, βαρύνονται με πολλά προβλήματα. Οι συστάσει όμω τη έκθεση θα αποτελέσουν βάση για μελλοντικέ εργασίε. Ένα σχόλιο όμω, θέλω να κάνω και αυτό αφορά το κοινωνικό ντάμπινγκ. Όλοι τελευταία μιλούν γι' αυτό οι μεταφορείς και οι εργαζόμενοι των μεταφορών θα πρέπει να εργάζονται σε αξιοπρεπείς συνθήκες και να αμείβονται αξιοπρεπώς. Παρ' όλα αυτά, η, το, έννοια του κοινωνικού dumping δεν θα πρέπει να γίνει αφορμή προκειμένου να περιοριστεί η πρόσβαση άλλων χωρών στην αγορά μεταφορών της Ευρωπαϊκής γιατί έχουμε δει καταχρήσεις και παρατυπίες σε αυτό το ζήτημα. Θα πρέπει επίσης να παρακολουθούμε πολύ στενά την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας στον δομέα των μεταφορών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σεχνάλοβα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, εξωτερικοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον ε, εισηγητή και τους δύο εισηγητές για την εξαίρετη δουλειά τους. Όσοι εισηγήτρια της προηγούμενης εκθέσεως θα συμφωνήσω με τον κύριο Φαντανικάμπο ότι χρειάζεται μια εσωτερική αγορά των μεταφορών που να προάγει, που να αξιοποιεί όλα τα μέσα. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται τα δίκτυα, η διασύνδεση. Και χρειαζόμαστε και να αντιμετωπίσουμε τις δύο διαφορές που έχουμε τις σημαντικές διαφορές που έχουμε στις υποδομές μεταξύ των παλαιών και νέων κρατών μελών και των νέων κρατών μελών στο επίπεδο των υποδομών και των εξυγχρονισμών τους που πρέπει να βελτιωθεί. Επίσης η πρόσβαση στις δημόσιες μεταφορές έχει πολύ μεγάλη σημασία αναφέρεται, όπως αναφέρονται και οι κοινωνικές συνθήκες εργασίας. Θα ήθελα λοιπόν με όλα αυτά να υποστηρίξω την έκθεση. Σας ευχαριστώ. Uh, Σας ευχαριστώ. Η κυρία Τζιλ Σέιμορ, ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Στην έκθεση ο εισηγητής προτείνει την εισαγωγή ε, τροχιοδρόμων, τροχιοδρόμων καλύτερα για τη βελτίωση των ε, μεταφορών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο κάτι τέτοιο κοστίζει 60 δισεκατομμύρια με 6 δισεκατομμύρια κόστος για τον πρώτο χρόνο. Με μειωμένο όμως ε, τον αριθμό των ε, επιβατών δεν νομίζουμε ότι αξίζει επένδυση. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια οδηγία η οποία δεν έχει φέρει αποτελέσματα και ανησυχώ ιδιαίτερα για την εσωπρόσθεσμη αυτή αξιολόγηση η οποία θα επέτρεπε θα απέτρεπε τα κράτη να περιορίσουν κάποιες ρυθμίσεις. Η έκθεση καλεί την Επιτροπή και την υποστηρίζει στην επιβολή μέτρων στα κράτη-μέλη για την επιβολή διοδίων για επιβατικά, επιβατικά και μικρά φορτηγά αυτοκίνητα. Αυτό ξεπερνά κάθε όριο. Ισχυρίζεται δε ότι μπορεί η Επιτροπή να ολοκληρώσει την ε, ε, δεύτερη φάση των ε, διευρωπαϊκών δικτύων των μεταφορών. Είναι παράδεκτη έκθεση και καλό συναδέλφους να την καταψηφίσουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Σαλίνη. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αίσθηση που μας δίνεται εξετάζοντας τη Λευκή Βιβλό και την έκθεση του συναδέλφου Βαντεγκάμπ είναι ότι έχει γίνει δουλειά διαμεσολάβησης και μάλιστα πάρα πολύ δύσκολη. Νομίζω ότι η Επίτροπος ε, μπορεί να το αναγνωρίσει και από τα όσα ακούσαμε να μας λέει βλέπουμε ότι υπάρχει εκτίμηση για μια πολύ λεπτό δουλειά ε, που ορισμένε φορέ προσπαθεί να διασκεδάσει τι απόψει των διαφόρων αντιπροσωπιών που έχουν τελείω διαφορετικέ θέσει. Κρίμα που στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύ συχνά συμβαίνει αυτό το οποίο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Σε έναν χώρο όπω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου θα μπορούσαμε στην πραγματικότητα να επιλύσουμε τις εντάσεις, ε, ελοχεύει ο κίνδυνο να φέρνουμε τι εντάσει τη κάθε χώρας. Ε, είναι λυπηρό αυτό. Ε, εγώ θεωρώ ότι η έκθεση θα πρέπει να υποστηριχθεί πλήρως. Ενδιαφέρεται κυρίω για τα θέματα που μα αποσχολούν, Παραδείγματο χάρη σε μένα αφορούν ιδιαίτερα οι σειροδρομικές μεταφορές και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία τα οποία μα επιτρέπουν να κατανοήσουμε πώ πώς μπορούμε να επενδύσουμε στις μεταφορές χωρίς να χρειάζεται να υλοποιούμε καπρίτσια τα οποία δεν θα έπρεπε να κάνει η Ευρώπη ε, για θέματα για τα οποία είμαστε ήδη πολύ αποτελεσματικοί. Υπάρχει δυνατότητα λοιπόν να έχουμε πολύ σημαντικές επενδύσεις που σέβονται και το περιβάλλον και η δυνατότητα που έχει αυτή η έκθεση να ευνοήσει αυτή την πορεία προς χρήσιμε επενδύσεις για την κινητικότητα των εμπορευμάτων και την κινητικότητα των ανθρώπων μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι και μέσω της πολιτικής μεταφορών η Ευρωπαϊκή Ήπειρος θα έχει την ανάπτυξη που της αξίζει. Ε, Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σαλίνη. Η Άγνες Ιουγκέριος. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι άρρωστοι πιλότοι που παρόλα αυτά θέλουν ε, να πετάξουν, οι οδηγοί φορτηγών που πρέπει να ε, οδηγούν 24 ώρες το 24ωρο γιατί φοβούνται να χάσουν τη θέση εργασίας τους. Νέοι ναι, άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να σεβαστούν τους κανόνες ε, διότι ξέρουν ότι δεν θα τους πιάσει κανείς ε, είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να αποδεχτούμε. Η πρόταση της έκθεσης αυτής είναι πάρα πολύ καλή και πρέπει να πω ότι χαίρομαι που επιτέλους οι χριστιανοδημοκράτες έχουν πιστεί ότι κάτι πρέπει να γίνει. Τα συγχαρητήριά μου λοιπόν κύριε Βαντεκάμπ. Τώρα πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει επιτέλους να δράσει. Η Επίτροπος εξέφρασε εδώ τις πολιτικές της επιθυμίες. Θεωρώ ότι είναι και η ώρα να επιδείξουμε φιλοδοξία για να υλοποιήσουμε συγκεκριμένα μέτρα ώστε να λήξει επιτέλους το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το τομέας αυτός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Ζορζ Μπάς τώρα για 1,5 λεπτό. Παρακαλώ. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να εκφράσω ιδιαίτερο τις ευχαριστίες μου προς τον συντονιστή μας κύριο Φαντερκάμπ, ο οποίος μπόρεσε, μέσα σε μπόρεσε να προτείνει βράχη μέσο και μακροπρόθεσμα μέτρα. Θα επικεντρωθώ σε δύο μόνο σημεία, μια και δεν έχω χρόνο. Καταρχάς τις οδικές μεταφορές. Γνωρίζουμε τα προβλήματα και τις προκλήσεις εδώ και πολύ καιρό ιδιαίτερα στο μέα της ασφάλειας, τα κοινωνικά, το περιβάλλον, τον ανταγωνισμό, δεν χρειάζεται νέα νομοθεσία. Στη συνεργασία με τα κράτη-μέλη χρειάζεται καλύτερη και αρμονική, κοινή υλοποίηση και ενισχυμένη έλεγχη. Μια υπηρεσία, ένας, ε, μια κοινή υπηρεσία θα ήταν ο κατάλληλος τόπος για να συναντηθούν αυτές οι αρμοδιότητες. Εδώ θα πρέπει να σημειώσω επίση για του σιδηροδρόμους ότι έχουμε φτάσει πια στο τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο. Ύστερα από 20 χρόνια προσπαθούμε να δώσουμε πλέον το ρόλο που αξίζει ο σιδηροδρόμους στι ενέργειε μεταφορέ. Ε, έναντι των ενέργειων μεταφορών υπάρχει κίνδυνο οι σιδηροδρόμοι να χάσουν όλο και περισσότερο έδαφο ανταγωνιστικά και πρέπει να δοθούν ε, ε, σαφεί λύσει. Κύριε Επίτροπε, εσείς ύστερα από χρόνια στασιμότητας ε, των προηγούμενων, των προκατόχων σας, έχετε πλέον να αναλάβετε μέτρα που θα ενισχύσουν και την, ε, τον οικονομικό κλάδο των μεταφορών και θα βελτιώσουν την ε, ανταγωνιστικότητά τους και τις θέσεις εργασίας για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και τώρα η κυρία Κλούνα. Ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ, Επιτροπέ. Ευχαριστώ τον κύριο Καπ, τον εισηγητή, για τις προσπάθειες του. Ε, προσπάθησε να καταλήξουμε σε ένα ισόρροπο κείμενο συμβιβαστικό και ελπίζω ότι θα υπερψηφιστεί αύριο. υπογραμμίζει τη, συμφωνία των μετα... την, ε, τη σημασία των μεταφορών για τη σύνδεση των περιφερειακών περιοχών, δημιουργία θέσεων της κλπ. Αλλά στο κέντρο της πολιτικής και των υπηρεσιών μεταφορών θα πρέπει να είναι ο επιβάτης, αλλά και οι επιχειρήσεις, γιατί και αυτές εξαρτώνται πάρα πολύ από τις ε, υποδομές μεταφορών. Ε, σε ό,τι διάφορα τι ενέργειες μεταφορέ, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι οι μεταφορείς ε, ανταγωνίζονται πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο, σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Ο κόσμος μικραίνει και πάει. Οι επιβάτες μετακινούνται πολύ εκτός Ευρώπης πια. Ασία, Αμερική, Αυστραλία, οπότε και οι αερομεταφορείς θα πρέπει να ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Και θα πρέπει να το δούμε πώς μπορεί να υποστηριχθεί αυτό. Πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που εμποδίζει τους αερομεταφορείς μας και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον ανταγωνισμό. Ευχαριστώ. Τώρα περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Ο λόγος... Στην Κλάουδια Μοντέρο Αγκιάρ. Ευχαριστώ. Είμαστε ακόμα μακριά από την ε, επιτεύξη ενός ε, νέου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών, αλλά ξεκινάμε να κινούμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση. Γι' αυτό το λόγο η εργασία του εισηγητή και των σχεδόν εισηγητών είναι πολύ θετική. Ε, γίνονται αναφορές στις θαλάσσιες μεταφορές και στην ανάγκη να βελτιώσουμε τη, τους λιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν χωρίς καθυστέρηση να υποβληθούν προτάσεις για μέτρα για τη δημιουργία ε, λεωφόρων στη θα... θαλάσσιων λεωφόρων. Ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την άποψη των διεθνών θαλάσσιων οργανισμών ε, έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη τις, τις αρνητικές επιπτώσεις θα μπορούσαν να έχουν ε, να έχει ανάπτυξη, ε, μια συγκεκριμένη ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών στα ε, νησιά μας. Θα πρέπει να, ληφθούν, να υπόψη ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των επιδράσεων στις, στις θαλάσσιες Ευρωπαϊκής, νησιωτικές περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλώ πολύ να τηρείτε το χρόνο σας, γιατί αλλιώς θα πρέπει να σας διακόπτω. Κυρία Άντρισον. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται για μια έκθεση πνοής με πολύ σοβαρές προτάσεις, ιδιαίτερα την ανάγκη για τη ρυθμίση των, πολλέ, των λιμένων, το ζήτημα των πολύ μεγάλων φορτηγών, το ζήτημα των σιδηροδρόμων. Στα, στις προτάσεις αυτές, ε, λείπουμε που θα πω, θα καταψηφίσουμε η εργατική της Βρετανίας. Ωστόσο υπάρχουν άλλα σημεία θετικά, όπως σε παραδείγμα η μείωση κατά 60% στο 2050 των εκπομπών ε, αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές εν της διασκέψης των Παρισίων. Είναι πάρα πολύ σημαντική η δεσμεύση αυτή και θα ήθελα ιδιαίτερα να τονίσω την ανάγκη για επενδύσει στον τομέα των μεταφορών. Οι επενδύσει μεταφορέ στο Λονδίνο, την ιδιαίτερη μου πατρίδα, δεν παρακολουθεί τι ανάγκε του όλο και αυξανόμενου πληθυσμού. Το ίδιο ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν κατεπηγόντω να δώσουμε απαντήσει στα ζητήματα αυτά, στα μεγάλα αυτά κενά που έχουμε και ε, με επιμονή τα επόμενα χρόνια να προχωρήσουμε, να αναγνωρίζοντα βεβαίω ότι έχει ρόλο και ο ιδιωτικό τομέα, αλλά πρέπει να δώσουμε την έμφαση στι δημόσιε επενδύσει και τι μεταφορέ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Νότη Μαριά έχει το λόγο. Οι μεταφορέ είναι καθοριστική σημασία για την οικονομική ανάπτυξη τη Ευρώπη. Η αναβάθμισή του πρέπει να γίνεται με γνώμονα τον επιβάτη και την προστασία του περιβάλλοντο. Οι μεταφορέ όμω ευθύνονται για το 25% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι ο δεύτερος σε μέγεθος τομέας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά τον τομέα της ενέργειας. για τον λόγο αυτό πρέπει η ευρωπαϊκή ένωση να προωθήσει τις εναλλακτικές μεταφορές να προωθήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ιδίως τους σιδηροδρόμους. στον τομέα των οδικών μεταφορών πρέπει να ενισχυθούν οι υποδομές προκειμένου να έχουμε μείωση των οδικών ατυχημάτων αλλά και να υπάρξουν ενισχυμένοι έλεγχοι ταυτόχρονα η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να ενισχύσει τις θαλάσσιες μεταφορές προκειμένου οι κάτοικοι των νησιωτικών περιοχών και ιδίως του αιγαίου να έχουν συνεχή πρόσβαση στην ενδοχώρα. ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Η κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίκα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την Επίτροπο και ευχαριστώ και τον εισηγητή για τις προσπάθειές του. Η Ευρώπη χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα κινητικότητας διαλειτουργικής που θα βελτιώνει και τη βιωσιμότητα από πλευράς περιβάλλοντος αλλά και για τις ίδιες τις μεταφορές. Ε, οι μεταφορές είναι το 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και το γεγονός ότι υπάρχουν συγκεκριμένα συμφέροντα είναι ο λόγος για τον οποίο δεν τηρούνται αρκετές ευρωπαϊκές νομοθεσίες που αν εφαρμόζοντας θα βελτίωναν την οικονομία όλων. Πρέπει να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις ε, με βάση όσα έχουν συμφωνηθεί και ε, να υπάρχει προστιθέμενη αξία για όλο το σύστημα. Πρέπει να σκεφτούμε όλους τους χρήστες και αυτούς που έχουν προβλήματα κινητικότητας ε, όταν ασχολούμαστε με τα δικαιώματα των επιβατών. Θα πρέπει να έχουμε την ηγετική θέση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας στις μεταφορές το μέλλον της οικονομίας μας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας είναι αυτό το οποίο θα βελτιώσουν τις δυνατότητες που έχουμε και κυρίως θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και την κλιματική αλλαγή. Ευχαριστώ πολύ. Η Κατρίνα Κονέτσνα τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον Ισηλιό, συντονίστρια της Αρμόδιας Επιτροπής. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερα που ενεργειακή πολιτική λαμβάνεται υπόψη στον τομέα των μεταφορών. Πρέπει να χρησιμοποιούμε καλύτερα τους πόρους σε όλα τα συστήματα μεταφορών, προκειμένου να διασφαλίσουμε καλύτερη χρήση των δυνατοτήτων που έχουμε. Όπως ε, είπε ο εισηγητής, ε, στους 10 στόχους της Λευκής Βίβλου δεν, υπάρχουν θέματα, δεν υπάρχουν θέματα ανάπτυξης κοινών μεταφορών που θα μειώσουν ε, την επιβάρυνση από τις εκπομπές για το περιβάλλον. Θα πρέπει να υπάρχει μια κινητικότητα και για τους ποδηλάτες αλλά και για τους ηλικιωμένους. Είναι θέματα στα οποία θα πρέπει να επενδύσουμε. Είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι οι θετικές συνέπειες αυτών των επενδύσεων θα βοηθήσουν ε, όλα τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη επένδυση σε υποδομές ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε τις σιδηροδρομικές μεταφορές, τα διευρωπαϊκά δίκτυα και τη διασύνδεση στην Ευρώπη. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης στα δίκτυα αυτά. Ο κύριος Κόχα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για ένα λεπτό. Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Οι μεταφορέ ε, επηρεάζουν την καθημερινή μα ζωή. Δεν πρόκειται για την οικονομία, το περιβάλλον, ε, τι κοινωνικέ πτυχέ, ε, τον τουρισμό, την κλιματική αλλαγή και όμως ε, δεν, του δίνουμε, δεν τους δίνουμε την απαραίτητη σημασία. Έχουν πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν για την ποιότητα ζωής και στο μέλλον των πολιτών μας οι μεταφορές. Αυτή η καταγραφή λοιπόν της κατάστασης και η στροφή προς ε, μια καλύτερη κινητικότητα ε, τη εκθέσεω έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και ευχαριστώ τον κύριο Φαντανικάμπ. Νομίζω ότι θα πρέπει ωστόσο να κοιτάξουμε πιο προσεκτικά και άλλα σημεία, όπω ε, ε, την εμβαλωματική εικόνα παρουσίαση στο σύστημα των διοδίων στην Ευρώπη, το ζήτημα τη οδική ασφάλεια που θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία όπως άλλωστε καταγράφεται και στην έκθεση, αλλά και χρειάζονται συγκεκριμένοι στόχοι, μια στρατηγική για το περιορισμό του αριθμού των ε, ε, βαριών τραυματισμών στην Ευρώπη και ιδιαίτερα άνωτατο επίπεδο για την ε, ε, αλκοολεμία στην Ευρώπη. Σου οδηγού, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία Γιάρα Σέντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτέλους ο εισηγητής για μια φορά μας υπέβαλε μια συνολική εικόνα του μεταφρόνου στο μέλλον. Ε, πρώτο θέμα όμως η οδική ασφάλεια. Έχουν αυξηθεί τα, θέματα, τα θύματα, ε, έχουμε χάσει τη μάχη. Η κρίση χειροτερεύει και τις υποδομές και τα οχήματα και περιμένουμε προτάσεις από την, από την Επίτροπο. Ε, η ασφάλεια τώρα εναντίον τη της τρομοκρατίας ε, στην ε, Μαδρίτη αλλά και στο Λονδίνο και στο Παρίσι έχουν γίνει σε μεταφορικά μέσα τρομοκρατικά χτυπήματα περιμένουμε ότι το Συμβούλιο θα κάνει προτάσεις και γι' αυτό η αντίστοιχη ομάδα η όρια των εργαζομένων η υγεία τους είναι πολύ σημαντική επίσης για ποιο λόγο οι νέοι βρίσκονται σε ανεργία ενώ τα μεταφορικά μας ε, μέσα δεν μπορούν να βρουν πληρώματα και υπαλλήλου για την ε, αλλαγή της κοιτάλης σε νέα γενιά. Η βιωσιμότητα. Σε ό,τι αφορά την αστική κινητικότητα θα πρέπει να στηρίξουμε τη χρήση των ε, ποδηλάτων και το τραμ. Επίσης χρειαζόμαστε αυξημένο προϋπολογισμό ε, και το Ταμείο Στατικών Επενδύσεων σίγουρα θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί επιπλέον ε, για να ενισχύσει τον μηχανισμό συνδέοντας την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Gracias. finally, on behalf of Η ε, κυρία Επιτροπός έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για τα πολύ χρήσιμα και συγκεκριμένα σχόλια σας. Τα σημειώσαμε όλα. Οι παρατηρήσεις σας και η εκθεσή σας θα ληφθούν υπόψη στην ε, ολοκλήρωση της έκθεσης εφαρμής Λευκής Βίβλου, την οποία θα τελειώσουμε μέχρι το τέλος του χρόνου. ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό που όλοι αναγνωρίζουμε τη σημασία των μεταφορών για την άπτυξη, την απασχόληση και για το συνολικό διεθνή ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πω δύο λόγια καταρχήν για τη διαδικασία. Η δημόσια διαβούλευση, η διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους ε, ολοκληρώθηκε με πολλά από τα εφαρμοστικά μέτρα της Λευκής Βίβλου του 2011 ε, έχουν υλοποιηθεί πρόσφατα οπότε δεν είναι δυνατόν να γίνει πλήρης αξιολόγηση της Λευκής Βίβλου. Θα αξιολογήσουμε ότι έχει ήδη εφαρμοστεί. Ε, και θα δούμε τι έχει γίνει πλέον απαρχαιωμένο, τι έχει ξεπεραστεί και τι απομένει να γίνει. το πολιτικό και το οικονομικό πανόραμα βέβαια έχει αλλάξει μεταξύ, αλλά από ό,τι φαίνεται οι βασικές διατάξεις της Λευκής Βίβλου παραμένουν επίκαιρες και αξίζουν να υλοποιηθούν. Κατανοώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνεί με αυτή την προσέγγιση. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω μια ακόμα φορά τον κύριο Βαντερκάμπ και όλο το Κοινοβούλιο που αποφάσισε να λάβει αυτή την πρωτοβουλία. Όπως ανέφερα και στην εισαγωγή μου, συμφωνούμε με τις, ε, σε ό,τι αφορά τις ε, βασικές γραμμές για το μέλλον. Κα, ε, ακούω διάφορες εκκλήσεις για δράση και μου αρέσει αυτό. Ας συνεργαστούμε για τις πρωτοβουλίες οι οποίες πραγματικά θα μας βοηθήσουν να σημειώσουμε πρόοδο. Ευχαριστώ. Και τώρα ο λόγος στον συγητή τον κύριο Βιν Βαντενκάμπ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω την Επίτροπο και τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους, ακόμα και για τις επικρίσεις. Η κυρία Φώστερ έφυγε δυστυχώς, αλλά εγώ την κατανοώ απολύτως και λογικά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το λάβουμε υπόψη στην περαιτέρω υλοποίηση. Κύριο ε, Πρόεδρε, η μεγάλη πρόκληση είναι ότι αυτή η λευκή βίβλος και ενδιάμεση αναθεώρηση ε, είναι να μην μείνει κενό γράμμα. Θα πρέπει να υλοποιηθεί και θα πρέπει τα επόμενα χρόνια να δούμε πώς μπορούμε να ελέγξουμε ότι θα εφαρμοστούν αυτά τα οποία επισημάναμε ε, και που θα εγκριθούν αύριο θα πρέπει να υπάρχει κάποιο σημείο ισορροπίας. Να μην υπάρχουν τόσοι πολλοί κανόνες, αλλά μεγαλύτερη βιωσιμότητα, μεγαλύτερες δυνατότητες να έχουμε ωφέλη και να μην ξεχνούμε και τις κοινωνικές πτυχές. Όλα αυτά θα πρέπει κάπως να τα πλαισιώσουμε και αυτό ε, θα είναι και επιτυχία για την Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, θα μπορέσουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για τις μεταφορές με αυτά τα λίγα πράγματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.